Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Προηγουμένως, θέλω να θυμίσω μόνο ότι σήμερα έχουμε και ε, παθητικά φιλανδικά, δηλαδή ε, μπορείτε να μιλάτε φιλανδικά, αλλά όχι να ακούτε φιλανδικά. Θα δώσω μέσω στο λόγο στον κύριο Πάβο Βάιρινεν, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης για να μας κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Λαβία. Και καλησπέρα σας, συνάδελφοι. Τη Επιτροπή Περιβάλλοντος, τη Επιτροπή Γεωργίας και τη Επιτροπή Ανάπτυξης και των τριών επιτροπών. Καλωσορίζω θερμά την κυρία Αγκοστίνη εκ μέρους του ΦΑΟ και όλους εκείνους που μας παρακολουθούν για αυτό το σημαντικό ε, θέμα το οποίο δεν έχει πάντα την προσοχή που του αξίζει. Θα ήθελα καταρχάς να σας διαβιβάσω ε, ε, τις ένα μήνυμα και τη συγγνώμη της κυρίας Μακαβάν της Πρόεδρου της Επιτροπής μας, που κολλείεται και δεν παρευρίσκεται. Αλλά στο χρήμα πρέπει να αλλάξει λοιπόν και η διατροφή και η γεωργία. Και αυτό είναι το θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας διατροφής. Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο ΦΑΟ, πώς ε, η διατροφή και η γεωργία πρέπει να αλλάξουν στα πλαίσια της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και τι μπορούμε για να, να, να κάνουμε για να διευκολύνουμε αυτή την αλλαγή. Γνωρίζετε ότι περίπου 800 άτομα, εκατομμύρια άτομα ε, υποφέρουν από χρόνια πείνα και υποσυτισμό. Και στόχος μας είναι μέχρι το 2030 να έχει εξαλειφθεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει όμως για να εξαλειφθεί η πείνα να γίνουν πολλά, όχι μόνο λόγια, αλλά έργα και μάλιστα αποτελέσματα που να διαρκούν θα πρέπει να αυξήσουμε τη σοδιά μας, γιατί αυξάνεται και ο παγκόσμιο πληθυσμό και θα πρέπει να μπορούν να τρέφονται οι πληθυσμοί της γης από την παραγωγή της γης. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να γίνει αυτό με βιώσιμο τρόπο. Όχι τόσο με τη βιομηχανική γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο, την εντατική, όπως έχει γίνει σε πολλά μέρη του κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά αυξάνοντας την παραγωγικότητα της μικρής γεωργίας, των μικρών γεωργών που παράγουν πάνω από 70% ήδη των παγκοσμίων τροφίμων, αλλά συχνά μόνο σε επίπεδο επιβίωσης. Είναι τεράστια δυνατότητα να παράγουμε περισσότερα αν αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των μικρών αγροτών σε ό,τι αφορά τα εφόδια, τις υπηρεσίες, η πρόσβαση σε αυτές, πρόσβαση σε νερό, σε γέες και σε πολλές χώρες είναι πολύ σημαντικό να έχουν και την ε, σωματική τους ακαιρεότητα δεδομένη, να υπάρχει ασφάλεια δηλαδή στη χώρα. Επίσης οι μέθοδοι παραγωγής θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και στις προκλήσεις. Πρόσβαση σε ενημέρωση επίσης για μικρούς ενδιαφερομένου, ε, μικρούς αγρότες ε, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Χάρη στα κινητά τηλέφωνα μπορούν οι μικροί ε, αγρότες να ενημερώνονται ας πούμε για τις μετεωρολογικές συνθήκες, για τον καιρό, για τις διακοιμάσεις των τιμών των προϊόντων που παράγουν και των καλλιεργειών τους. Στο τσάντ για παράδειγμα, που ο παγκοσμίος είναι δεύτερη σε πείνα, δεν έχουν μετρολογική υπηρεσία ε, που να προβλέπει τον καιρό. Βλέπουμε ότι χρειάζονται υποδομές και στις πιο φτωχές χώρες. Η κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερη πρόκληση ε, για την ε, επιστημιστική ασφάλεια. Πάνω από 70% των φτωχών αυτού του κόσμου εξαρτώνται από τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους για την ίδια τους την επιβίωση. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ε, περιβαλλοντικές συνθήκες που αλλάζουν και σε ακραία ε, καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες, όπως είναι η επέκταση των ε, ερήμων και η αποψήλωση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις και να μπορούν πιο, να είναι πιο ανθεκτικοί οι πληθυσμοί της υπαίθρου στις κλιματικές αλλαγές και αδειξότητες, ε, χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Να σας εξηγήσω λίγο τι κάνει το Κοινοβούλιο. Στην τελευταία εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, εγκρίναμε ένα ψήφισμα ε, για τους παγκόσμιους στόχους και τις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστημιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Η έκθεση ήταν της δικής μας Επιτροπής, ΔΕΒΕ. Το Κοινοβούλιο εδώ υπογράμμισε τη σημασία προώθησης ε, συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της ε, πείνας και του υποσυτισμού, ιδιαίτερα των παιδιών και μάλιστα κατά τις πρώτες χίλιες ημέρες της ζωής τους. Ε, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ε, δεσμεύσει μας και επιπλέον ένα δισεκατομμύριο ευρώ δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή για να φτάσουμε στους στόχους ε, του ΟΗΕ και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης για να τερματιστεί ο ποσιτισμός και η φτώχεια μέχρι το 2030. Ε, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων τις δυνατότητες για αύξηση της παραγωγικότητας των μικροκαλλιεργητών με γεωργικά συστήματα και συστήματα διατροφικά που να ανθίστανται στα καιρικά φαινόμενα και να μπορούν να τρέφουν το πληθυσμό ε, της γης που θα είναι 8,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον και την βιοπικιλότητα. Η ε, απόφαση του Κοινοβουλίου και τα ψηφίσματα ε, θέλουν να υποστηρίξουν τους μικρούς αγρότες πάντα ε, με νέες γεωργικές πρακτικές, πιο παραγωγικές, πιο ανθεκτικές ε, και πιο ευφυείς σε σχέση με το κλίμα. Αγροοικολογικές δηλαδή, χρηστές πρακτικές έτσι ώστε να σταματήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος και να βελτιωθεί η απόδοση ε, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βελτιωθεί και η διατροφή. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι έχει σημασία να ενέχονται πρόσωπα, ε, συνεταιρισμοί, εταιρείε, όλοι ενεχόμενοι στη Γεωργία, ε, για να βρούμε λύσεις καινοτόμες για τις βέλτιστες γεωργικές πρακτικές και συστήματα που να μπορούν να τρέφουν ε, τον πληθυσμό σε ένα κόσμο που αλλάζει. Τις τελευταίες δεκαετίες αναλάβαμε σημαντικές δεσμεύσεις κατά πολέμησης κλιματικής αλλαγής και πρόθεσης της αντίστασης της γεωργίας. Στη Ρώμη έγινε το 1996 η πρώτη σύνοδος κορυφής και πιο πρόσφατα έχουμε τη Συμφωνία του Παρίσιου πέρσι και τους ε, στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί και μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, στρατευτεί σε αυτή την πορεία με φιλοδοξία για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και η ε, καταστροφή του περιβάλλοντος. Έχουμε μεγάλη ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθούμε ε, στις υποχρεώσεις μας και να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αρχίζουμε με αυτό το μήνυμα μέσω βίντεο από τον κύριο Όγκρατ, και τον Ευρωπαϊκό Γραμματέα του Οργανισμού Επιστημισμού και Γεωργία των Ηνωμένων Εθνών ΦΑΟ. Ladies Κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί φίλοι, φέτος η Παγκόσμια ημέρα για τη διατροφή έχει αφοσιωθεί στο και αφιερωθεί στο να αναλυθεί πώς η γεωργία και η διατροφή μπορούν να βοηθήσουν τόσο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, ε, συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Γιατί βλέπουμε ότι έχει γίνει α, ακανόνιστο και, άτακτο το τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται ο καιρό και έχουν ε, αυξηθεί η ασθένεια όπως επίσης ε, και ό,τι επηρεάζει την παραγωγικότητα της γεωργίας και αυτό επιδρά στην ε, διατροφική ασφάλεια. Και όπως πάντα οι πιο φτωχοί, οι πιο πεινασμένοι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο, το 80% εξ αυτών ζουν στην Ήπεθρο και βγάζουν το προστοζήν για να θρέψουν τις οικογένειές τους ακριβώς από τον ε, κλάδο ο οποίος βίσταται περισσότερο αυτές τις επιπτώσεις. Οπότε βλέπουμε ότι η αλλαγή του κλίματος υπονομεύει τις ε, προσπάθειες ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την ε, πείνα και τις άλλες μορφές υποσυτισμού μέχρι το έτος 2030 περίπου 800 εκατομμύρια είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ασφάλεια σε σχέση με την διατροφή, των επισητισμό τους περίπου 160 εκατομμύρια ανήλικοι κάτω από την ηλικία των 5 ετών έχουν πληγεί από αυτό το φαινόμενο και υπάρχει όλο ένα και περισσότερη συνειδητοποίηση ότι η γεωργία μπορεί να βοηθήσει στον μετασχηματισμό και να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές του κλίματος. Οι δράσεις ούτω ώστε να είναι πιο ανθεκτική η γεωργία είναι κάτι πάνω από τη μείωση των επιδόσεων και πέρα από την απλή προσαρμογή, γιατί ακριβώς εμείς θέλουμε να φέρουμε την ε, ε, προσαρμογή, αλλά επίσης και να συγκρατήσουμε τις επιπτώσεις αλλαγής του κλίματος, οπότε αυτή η μέρα της διατροφής ε, το 2016 είναι μια ευκαιρία ούτως ώστε να δούμε πώς καλύτερα θα ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Στο COP21 του Δεκεμβρίου, στο Παρίσι, περισσότερες χώρες ε, κάλυψαν και τη γεωργία στις ε, εθνικές ε, καθορισμένες συμβολές. Και τον Νοέμβριο αυτές οι χώρες πρόκειται να συνέλθουν στην ΚΟΠ 22 του Μαρόκου, ούτω ώστε να μπορέσουν να κινητοποιηθούν και να δεσμευθούν. Οπότε με τη συνεργασία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της γεωργίας για τον μετασχηματισμό. Αλλάζει το κλίμα, αλλά πρέπει να αλλάξει και η γεωργία, όπως επίσης και η διατροφή. Ευχαριστούμε κύριε Ντασίλβα για τα όσα μας είπατε και τώρα η σκητάλη στην κυρία Αστρίντ Αγκοστίνη που είναι ανώτερη υπάλληλο όσον αφορά του φυσικού πόρου στην Διεύθυνση για την Αλλαγή του Κλίματο και των περιβάλλων τη ε, οργάνωσης για τη γεωργία και τη διατροφή του ΟΗΕ, της ΦΑΟ. Εκτός μικροφώνου η κυρία Αγκοστίνη. Αγαπητοί πρόεδροι της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επιτροπής Γεωργίας, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τις δύο Επιτροπή σα μου είναι αυτή την ε, ευκαιρία. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Παγκόσμια ημέρα για την διατροφή ε, γιορτάζεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε τι έχουμε να αναδείξουμε με αυτή την ευκαιρία. Τόσο να υπάρξει περισσότερη διατροφική ασφάλεια. Να δούμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε τάξει. Ποια είναι η μεγάλη πρόκληση, είναι η διατροφική ασφάλεια στα πλαίσια του μεταβαλλουμένου κλίματος. Θα πρέπει να διαθρέψει περισσότερο τώρα η, η γεωργία. Η αλλαγή του κλίματος είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την επιτεύξη αυτού του στόχου. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν και η αλλαγή του κλίματος πλήσει πολλές εμπισόμενες χώρες. 22% της συνολικής ε, ζημίας υφίσταται η γεωργία. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι η γεωργική παραγωγή μειώνεται από 10-25% και αυτό ίσως ε, αυξηθεί με το 2050. Όσον αφορά δε την αλία στις τροπικές περιοχές, η μείωση μπορεί να φτάνει το 40 με 60%. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα με το έδαφος, το 1 τρίτον του εδάφους έχει υποστεί χειροτέρευση. Επίσης, οι διάφορες ασθένειες και μολύνσεις ε, είναι κάτι το οποίο εξαπλώνεται αυτές που αφορούν τα φυτά. Οπότε βλέπουμε ότι η γεωργία δεν είναι θύμα μόνο της κλιματικής αλλαγής. Πλήσεται και από τις εκπομπές τις σχετικές με το φαινόμενο θερμοκηπίου. Να, βλέπετε τι γίνεται εδώ με τα δάση και τις λοιπές χρήσεις της γης. Η καταστροφή των δασών, ε, η κτηνοτροφία, κακή διαχείριση του εδάφους. Και όπως και σε άλλους κλάδους, πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες για το πώς θα υπάρξει συγκράτηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλληλεγγύης του κλίματος. Εδώ μιλούμε για τον πρωτογενή τομέα και για το τι ζημία υπάρχει εκεί και τι πάει χαμένο από την παραγωγή τροφίμων. Η χρησιμοποίηση της ενέργειας και αυτή είναι ένας ε, παράγον που επηρεάζει. Είναι σημαντικό τώρα με αυτή την ευκαιρία να δούμε πόσο σημαντική είναι η γεωργία όσον αφορά το τι γίνεται αναχώρα και τι στρατηγικές έχουν εκπονηθεί από κάθε χώρα. Σε αυτές τις εθνικές συμβολές, τα INDC, που αποτέλεσαν φεμέλιο για τη Συμφωνία των Παρισίων, ε, αναδεικνύει το ρόλο της γεωργίας. Αυτά τα ε, INDC θα γίνουν NDC και πρόκειται έτσι να οργανωθεί η δράση κάθε χώρα σε σχέση με την του κλίματος. Παρασόν αφορά την συγκράτηση των ελληνικών συνεπειών, σχεδόν 90% όλων των χωρών ε, προσπαθούν να αναπτύξουν κάποιες δράσεις συγκράτηση των αρνητικών συμπιών μέσα από τη Γεωργία. Αυτό αφορά 86% των αναπτυσσομένων χωρών. Και αυτό αφορά επίση και τις ε, εκπομπές των ε, αερίων ε, θερμοκηπίου των σχετικών εκπομπών. Τώρα, όσον αφορά την προσαρμογή, εδώ είναι ακόμη πιο σημαντικό ο ρόλο τη γεωργία και βέβαια δεν καλύπτονται όλα τα INDC. Αυτό δεν ήταν μέσα στις βασικές προϋποθέσεις της συμφωνίας. Αλλά εδώ έχουμε τέτοια μνήμα της προσαρμογής που επίσης έχει σχέση με τον τομέα της γεωργίας. Κάτι άλλο πιο σημαντικό. Όχι μόνο επομένως ή πρωταγωνιστικό ρόλο η γεωργία στην συγκράτηση των συμβίων και στην ε, προσαρμογή, αλλά είναι και οι συνέργειες που αφορούν την γεωργία. Οπότε και έτσι διαφοροποιείται η γεωργία από τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση πάντα με την αλλαγή του κλίματος. Περίπου 50 χώρες δίνουν προτεραιότητα σε κάποιες δράσεις που έχουν σχέση με αυτές τις συνέργειες. Περίπου 30 χώρες επίσης ε, χρησιμοποιούν την έννοια της ε, ευφυούς κλιματικά γεωργίας. Τι είναι αυτή η γεωργία, η κλιματικά εφής Η ΦΑΟ εισήγαγε το 2010 αυτόν τον όρο και ε, πολλοί συμμετέσχουν στο σχετικό προβληματισμό. Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία βοηθά για τη διαχείριση και αλλαγή στην γεωργία που να οδηγήσει σε διατροφική ασφάλεια υπό τις συνθήκες της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει να αυξηθεί η ε, παραγωγικότητα και τα εισοδήματα. Η, να είναι πιο ανθεκτική η γεωργία στην αλλαγή του κλίματος και ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βλαπτικές εκπομπές όπου είναι δυνατό. Να υπάρξουν συνέργειες και επίσης να γίνει διαχείριση των ε, αντισταθμιστικών συνεπειών όπου αυτές υπάρχουν. Τώρα, πάρα πολλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε τόπου. Δεν πρόκειται για κάποιες καθιερωμένες και καθορισμένες προοπτικές. Είναι οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει τους τρεις προανεφερέντες στόχους ε, κάθε φορά στη συγκυρία και στις συνθήκες που ισχύουν. Επομένως αυτό έχει κοινωνικό, οικονομικό περιεχόμενο και ισχύει ε, οριζόντια ή μάλλον ισχύει σε κάθε επίπεδο όπως τίθενται κάποιοι στόχοι από την κάθε χώρα καταβάλλεται προσπάθεια με συνέργειες να επιτεθούν αυτοί οι στόχοι είτε σε επίπεδο εκμετάλλευσης, είτε εθνικό, είτε περιφερειακό. Και είναι μια προσέγγιση για κάθε κλάδο και τομέα. Δεν αφορά μόνο την ε, γεωργία. Είναι και θέμα κοινωνικής προστασίας. Είναι και θέμα ασφάλισης. Και έτσι αναπτύσσεται αυτή η έξυπνη γεωργία. Επιτόπου τώρα. Ποια είναι η εικόνα που δίνει αυτού του είδους η γεωργία. Θέλουμε βιώσιμες πρακτικές, αλλά θέλουμε αυτό να γίνει με μακρόπνοη θεώρηση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα μακρόπνοα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος. Και υπάρχουν πολλές δυνατές προσεγγίσεις σε κάθε τομέα και υποτομέα. Αλλά δεν είναι μόνο το τι γίνεται σχετικά με την φτηνοτροφία, την γεωργία, την αλία. Είναι και θέμα διαφοροποίησης και έτσι να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν το εισόδημα. Για παράδειγμα, κοιτάξτε τι γίνεται με αυτόν τον ξηρό διάδρομο της Κεντρικής Αμερικής. Έχουμε κάποιο λοφόδες ε, τοπίο, κάποια βάλωτα εδάφια. Και εδώ Έχουμε κάποιες καινοτόμες λύσεις και κάποια συστήματα, οπότε τα δάση και η δασική γεωργία ε, καλύπτεται. Έχουμε κάποια δάση στις εκμεταλλεύσεις. Ποικιλία δέντρων και δέντρων που παράγουν φρούτα. Υπάρχει Υπάρχει επίσης διαχείριση βιολογικού υλικού. Για να δούμε τώρα. Η... αποτελέσματα ποια είναι. Αυξήση της παραγωγικότητας. Διαφοροποίηση στην παραγωγή όσον αφορά τις βασικές καλλιέργειες αλλά και τα δέντρα που παράγουν καρπούς. Μειώνουμε τη διάβρωση του εδάφους και εμπλουτίζουμε το έδαφος. Ε, ε, το, το έδαφος μπορεί έτσι να κατακρατήσει περισσότερο νερό, μείωση των κινδύνων και καλύτερη διαχείριση του τοπίου, του υδροφόρου ορίζοντα και των ε, εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα. Δεν πρόκειται μόνο για αυτές τις επιτόπου πρακτικές. Θα πρέπει να συνοδεύονται από διάφορες βάσεις πρώτα-πρώτα θα πρέπει να υπάρχει διαπίστωση του τι ωφελεί, τι είναι το πιο δόκιμο για την επίτευξη των στόχων. Άρα μέθοδος για να βρεθεί και να επισημανθεί η καλύτερη μέθοδος ή σύστημα και να μπορούν να επιλέξουν οι γεωργοί να στραφούν στο πιο αποδοτικό σύστημα. Και έτσι βρίσκονται νέε ισορροπίε και καλύτερα εισοδήματα με πιο βιώσιμε πρακτικέ. Τώρα, τι συμβάλλει σε αυτά η ΦΑΟ. κάποια δημόσια αγαθά και υποστήριξη σε κάθε χώρα. Δεδομένα, μεθόδους και μέσα ή εργαλεία. αναλύσεις ακριβώς όπως είπαμε προηγουμένως στην ε, παρουσίαση για το τι γίνεται με τα INDC. Κάποιοι κώδικες ιδεντολογίας, καθεντήριες γραμμές που αναπτύσσονται σε σχέση με το φόρουμ του ΦΑΟ. Επίσης, ανάπτυξη δυνατοτήτων για αυτές τις νέες μεθόδους και τα νέα εργαλεία ή μέσα. Διάλογος για την πολιτική που θα επιλεγεί. Για τη γεωργία, για το περιβάλλον και βέβαια παροχή συμβουλών και επικοινωνία. Όλα αυτά εν του COP22 τον Νοέμβριο. Εκεί η Γεωργία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και πρόκειται να εμπλακούν πάρα πολλοί από τους εταίρους μας. Συνεργασία θα γίνει και με την κυβέρνηση του Μαρόκου, ούτω ώστε να καλύψει η ΚΟΠ την Γεωργία και τους διάφορους υποτομείς της. Είναι μεγάλο αυτό το θεματολόγιο. Δεν είναι δυνατόν ένας μονοφορέας να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα χρειάζεται συνεννόηση και συνεργασία. Θα πρέπει να εξελίξουν πάντως ότι όλοι οι επιμέρους τομείς της γεωργίας ε, περιλαμβάνονται σε κάθε προβληματική για την αλλαγή του κλίματος. Και θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση σε σχέση με το κλίμα για την ε, γεωργία. Θα πρέπει να επίσης να υλοποιηθεί η αποφασιστήσα υποστήριξη στα εθνικά NDC. Και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, στόχου που έχει τάξει κάθε χώρα, αυτές τις προκλήσεις που έχουμε ε, επισημάνει. Α, επίσης θα πρέπει να σας τονίσω ότι μία έκθεση θα δημοσιοποιηθεί την Δευτέρα που θα αφορά την κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά την διατροφή, όσον αφορά την γεωργία. Για το εναλλαγή του κλίματος επίσης και όπως αναφέραμε προηγουμένως έχουμε δεδομένες τις εθνικές δεσμεύσεις, άρα είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για ανάληψη δράσης. Με αυτή την έκθεση λέμε ότι όσο καθυστερούμε τόσο περισσότερο ανεβαίνει το κόστος. Άρα τώρα που έχουμε την ευκαιρία ας ενεργήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Ζων Πιέρ Ολκίν της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ανάπτυξης ε, Γεωργής Ανάπτυξης ε, Καλό απόγευμα αξιότιμα μέλη αυτών των τριών επιτροπών. Είναι τιμή μου που μιλάω εδώ σήμερα. Καλωσορίζουμε και την έκθεση της ΦΑΟ που ε, ουσιαστικά συνάδει με τις δικές μας προσπάθειες. Θα σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες μας με τρεις λέξεις. Γνώση, χρήμα, πολιτικές. Προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στον τομέα της ε, έρευνας στην περιβαλλοντική πολιτική. Έξυπνη γεωργία, προσαρμογή, μετριασμός, ισορροπία μεταξύ των δύο. Όμως υπάρχει και ο αντίκτυπος. Η έρευνα που χρηματοδοτείται από χρήματα της ανάπτυξης πρέπει να έχει αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Δεν μας στάνουν κάποια βιβλία, κάποιοι τόμοι στη βιβλιοθήκη. Πρέπει η έρευνα που κάνουμε να έχει αντίκτυπο για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή είναι η ετήσια παρέμβασή μας στο σύστημα ECJR. Η έρευνα μας οδηγεί μετά στο ποιος μεταφράζει τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής στη γεωργία. Παραδοσιακά εμείς προσεγγίσουμε τις κυβερνήσεις για να το κάνουμε αυτό. Όμως ε, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι υπηρεσίες που παρέχουν τα τα κράτη ε, δεν είναι επαρκής. Τα χρήματα λοιπόν που ε, επενδύονται δεν αποφέρουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν και άλλες υπηρεσίες και άλλοι φορείς υπηρεσιών. Ο ιδιωτικός τομέας, ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες μεταξύ ευρωπαϊκών εταιριών και ξένων μπορεί να οδηγήσει στην μεταφορά των γνώσεων που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Οι ενώσει γεωργών τώρα. Οι ενώσει γεωργών μπορούν πραγματικά να επιφέρουν προσθέμενη αξία. Ε, αξία χρήσιμη για την έρευνα. Έρευνα η οποία είναι χρήσιμη για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Τώρα τα χρήματα. Ε, έχουμε και εδώ καινοτόμε ε, προσεγγίσεις. Καταρχήν έχουμε το AgriFi το παρουσίασε στην Expo του Μιλάνου τον Οκτώβρη πέρσι η Επίτροπος. Agrify είναι η γεωργική ε, χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έγινε για χρήματα ε, επενδύσεων κινδύνου για να μπορέσουν ε, να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις και να επενδύσουν στην έξυπνη γεωργία. Είναι δύσκολη η η προσπάθεια αυτή, διότι χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν πάνε εκεί που θέλουμε να πάνε, γιατί υπάρχει αυτό ο ρίσκο, αυτό ο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στι 24, Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Γιούγκερ ξεκίνησε το εξωτερικό σχέδιο επενδύσεων. Είναι ε, ουσιαστικά η ίδια αυτή προσέγγιση σε μεγαλύτερη κλίμακα μετά την ε, ατζέντα δράση τη Άντις Αμπέμπα ε, για να έχουμε πραγματικά μετρήσιμο αντίκτυπο στη ζωή εκατομμύριων. Θέλω να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σύντομα θα συζητήσει αυτή την πρόταση για το εξωτερικό σχέδιο επενδύσεων να εξετάξει το πολιτικό, να εξετάσει το πολιτικό σκέλος. Και τρίτον, οι πολιτικές. Εδώ έχουμε μακροσκελή συνεργασία με την ΦΑΟ, ε, έχουμε και μια ροή χρηματοδότησης προς τη ΦΑΟ, για να κάνουν πολιτικές για μας, μαζί μας, στις ε, χώρες εταίρους. Ήμουν πρέσβης και ξέρω ποια είναι η αξία ε, του λόγου της ΦΑΟ. Όταν δεν με άκουγε εμένα, ο εκπρόσωπος της ΦΑΟ είχε πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Εμείς όμως ερχόμαστε συμπληρωματικά ε, με το ΦΑΟ να πούμε ότι συνήθω η γεωργία και η έξυπνη γεωργία που έχει σχέση με την αλλαγή του κλίματος μπαίνει σε ζητήματα πολιτικά. Είχαμε πολλές κοινοδοτικές ερωτήσεις για το land grabbing. Είχαμε ένα πολιτικό παράγοντα ε, που είχε μια σειρά από προτερήματα, πλεονεκτήματα χάρη στη δράση του. Τώρα, μαζί με τη ΦΑΟ, τα καλύπτουμε όλα. Διακυβέρνηση, ζητήματα διαφθοράς, κράτος δικαίου, χρήση της γης, αλλά και συγκεκριμένες τεχνικές ε, συμβουλές για να μπορέσουμε όλοι να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση γεωργική, φιλική προς το κλίμα. Θα το δείτε και στη Μαρακές αυτό. Ε, η γεωργία δεν θα είναι πλέον κατηγορούμενος, θα παίζει ένα ρόλο και για την προσαρμογή αλλά και για το μετριασμό. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα συζήτηση με τους συναδέλφους. Ο πρώτος, ο Άλμπερτ Ντέστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α, αυτό το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας. Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεινάνε. Και είχα πει κάποτε στη Γερμανική Βουλή, αρκεί και 50% ε, των μέσων, των χρημάτων που δίνουμε για εξοπλισμούς, αν τα δίναμε στη Γεωργία, δεν θα πεινούσε κανείς αυτή τη γη. Και αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της Γεωργίας ή της κλιματικής αλλαγής, είναι μέγα πολιτικό πρόβλημα, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ταΐσει την ανθρωπότητα να έχει όλος ο, κόσμος ε, αρκετά τρόφιμα και οι πολιτικοί ηθήνοντες των χωρών αυτών φταίνε. Και πάλι συχνά μιλάω για τη Ζιμπάμπουε που ήταν ο Σιτοβολώνας στη Μεσημερινή Αφρική παλιά η Ροδεσία. Και τώρα ο κόσμος πεινάει. Αυτά είναι εγκλήματα. Ε, και δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Είναι πολιτική ευθύνη επιτόπου. Και ε, γεωργία και κλιματική αλλαγή. Την καθίζουν στο σκαμνί τη γεωργία. Θυμίζω όμως ότι πριν έρθουν οι Λευκοί στη Βόρεια Αμερική ε, είχαν ε, πολλά ζώα τα οποία δεν τα επηρέασαν οι κλιματικές αλλαγές. Ε, θα πρέπει να δίνουμε λοιπόν ε, ε, προγράμματα που να βοηθούν τους αγρότες, που να βοηθούν τους κτηνοτρόφους και ξέρουμε ότι από 800 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να τραφούν σωστά οι περισσότεροι είναι αγρότες. Ε, πήγα στη Βραζιλία ε, και σε ένα project βοηθήσαμε 500 οικογένειες για να μπορούν να έχουν αρκετό φαγητό με πάρα πολύ μικρό κόστος. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι μέτρα θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα τα αξιοποιήσουμε. και δεν έχει καμία σχέση η κλιματική αλλαγή σήμερα. Είχαμε και στο παρελθόν κλιματικές αλλαγές χωρίς εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα. Ας μην υπερβάλλουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα και να φροντίσουμε οι άνθρωποι αυτοί τα 800 εκατομμύρια να έχουν φαγητό και να μην τα φορτώνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανιώ κύριος Άγνιου. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν να στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όμως θα εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε ότι την περασμένη Πέμπτη 450 ευρωβουλευτές σε αυτό το σπίτι ε, ψήφισαν να μην έχουμε γάματα φόμικρων στην Ευρώπη. Ε, αυτοί οι 450 ε, ψήφισαν οι κατά, αλλά το τα γάματα φόμικρον είναι αυτά που θα μας σώσουν από την πείνα. Μπορεί να βοηθήσουν να αυξηθεί και η ποιότητα των τροφίμων που τρώμε. Παραδείγματο χάρη το χρυσό ρύζι στην Νοτιοανατολική Ασία. Επίσης ε, μπορεί να διαφυλάξει και την ποιότητα. Πρέπει λοιπόν με αυτή την τεχνική να οργώνουμε λιγότερο και να έχουμε έτσι καλύτερη ποιότητα γης. Ε, λοιπόν, λέτε ότι υπάρχει υπεθέρμανση λόγω των εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα. Θα μειωθεί, θα μειωθεί και θα μειωθούν και τα ρητά καύσιμα στη γεωρική παραγωγή με τα γάματα φόμικρον. Αν όμως ε, θεωρείτε ότι η, με την ε, ηλιακή ενέργεια ε, θα λύσουμε το θέμα, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι σε λίγο θα είναι πολύ πιο κρύος ο πλανήτης. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη η παραγωγή με κρύο κλίμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή όλα τα όπλα στη φαρέτρα μα και θα χρειαστούμε αυτέ τι νέε μεθόδου να το πω σε όλους. Ε, δεν πρόκειται να λύσετε τα, τα ε, αυριανά προβλήματα με χθεσινές μεθόδους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις στην αρχή της συνάντησης. Συμφωνώ ότι είναι ένα σημείο κλειδί στην προσπάθεια εκκλήρωσης της φτώχειας να χρησιμοποιήσουμε τη μοντέρνα τεχνολογία για να μπορέσουμε να δώσουμε τροφή σε αυτούς που πεινούν στον κόσμο. Εάν χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια για να εξασφαλίσουμε την παραγωγή τροφίμων, να χρησιμοποιήσουμε τη μοντέρνα τεχνολογία, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα χρήματα για να ταΐσουμε τους ανθρώπους και λιγότερο, λιγότερα χρήματα για να κάνουμε πολέμους. Έτσι θα υπήρχαν και λιγότεροι μετανάστες χωρίς τους πολέμους. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος δεν θέλω τώρα εδώ να προδικάσω το κατά πόσο ο πλανήτης θα είναι πιο ζεστός ή πιο κρύος στο μέλλον, αλλά η κλιματική αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στη γεωργία και αυτό αφορά και την Ευρώπη. μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα χρησιμοποιώντας όλα τα τρόφιμα που παράγουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει σπατάλη. Χρειαζόμαστε και δείκτες που να μας δώσουμε να καταλάβουμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Οι μέλισσες είναι ένας πολύ καλός δείκτης. Καλωσορίσαμε εδώ εκπροσώπους ε, της ΦΑΟ και θα ήθελα να πω ότι οι σλοβενικές ιδέες για την Διεθνή Μέρα ε, της Μέλισσας ε, σύντομα θα παρουσιαστούν και νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει για να ακολουθήσουμε ένα καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κυρία Ε, και ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι καλό που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα αλλά θα πρέπει να δούμε και την κατάσταση κατάματα, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Συχνά μιλάμε για το περιβάλλον, για τη φύση και τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Μα είναι πολύ σημαντική η γεωργία, ε, χωρίς εκπομπές ρήπων με, με ψηλή απόδοση. Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μετεγκατασταθεί η γεωργία και καλλιέργειες από την Ευρώπη αλλού. Δεύτερο, για το κόστος. Θα πρέπει να είμαστε ε, πραγματικά ε, συγκρατημένοι για τα ε, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και το κόστος και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό εξαρτάται και από την κτηνοτροφία και από την εκτατική κτηνοτροφία, τους βοσκοτόπους ε, και η Ευρώπη έχει μεγάλη καινοτομία ε, και οι οργανώσεις των γεωργών επίσης ε, πολύ συχνά και μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία. Μιλάμε συχνά για το μικρό αγρότη. Για πόσο καιρό είναι μικροί οι αγρότες μήπως να τους βοηθήσουμε να ενωθούν και να, μπορούν να παράγουν για να μην τους κατασπαράσουν όπως γίνεται στην Αφρική οι πολυεθνικές και η Κίνα. Εμείς ε, θα το χάσουμε αυτό το τρένο ή προλαβαίνουμε ακόμα. Ευχαριστώ κυρία Σανέρα Ροντρίγκεθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς ε, ε, εγώ μάλλον αυτή την ημέρα της διατροφής θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όταν μιλάμε για διατροφή πρέπει να έχουμε ως βάση το δικαίωμα των λαών να παράγουν τα βασικά τους τρόφιμα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τις ιδέες αυτές που ακούμε συνήθως να λένε ε, οι εκπρόσωποι των ε, θεσμών ότι η Ευρώπη πρέπει να παράγει για να, να θρέψει τον κόσμο. Όχι, η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την παραγωγή της και να επιτρέψει σε άλλες ε, περιοχές του κόσμου να παράγουν. Στο πλαίσιο αυτό, στο θέμα της παραγωγής τροφίμων, της εκρίζωσης, της φτώχειας, της καταπολέμησης, της κλιματικής αλλαγής, υπάρχουν σημαντικές πτυχές που πρέπει να έχουμε κατά νου η γεωργία στην Ήπεθρο, η βιογεωργία, η πρόσβαση στο νερό, η πρόσβαση στους σπόρους, πολύ σημαντικές πτυχές μαζί με τα μικρά κυκλώματα εμπορίας. Όταν όμως μιλάμε για τον, τον αριθμό των πεινασμένων στον κόσμο και όταν χρόνο με το χρόνο διαπιστώνουμε ότι αποτυχάνουμε, δεν φτάνουμε στους στόχους που θέτουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε όλο και πιο πολλούς πεινασμένους, φτωχούς, που δεν έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα. Να δώσω κάποια στοιχεία. Στην Ισπανία το 39% των παιδιών έχουν ε, προβλήματα διατροφής ή πεινούν και ένα σημαντικό ποσοστό είναι σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν πάμε λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντί να μπορέσουμε να εκριζώσουμε τη φτώχεια ανά τον κόσμο, με τις πολιτικές αυτές τις νεοφιλελεύθερες συνεισφέρουμε στο να αυξηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω από αυτό που είπε μόλις η Λίντια και ο κύριος Ντασίλβα ε, το είπε στο χαιρετισμό του στο βίντεο, αλλαγέ χρειαζόμαστε περισσότερο από στο παρελθόν. Ε, το τύχες Γιάννη τύχα πάντα δεν είναι επιλογή να συνεχίσουμε την ίδια τακτική. Στην Αφρική ε, μπορεί να υπάρχουν πολύ καλές ιδέες, αλλά στην πράξη ε, είναι πολύ διαφορετικές εξελίξεις από τις προθέσεις μας. Έχουμε αλλαγές ε, στην αντιμετώπιση των ζυζανίων και των ασθενειών. Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε και πάλι με χημικά φυτοφάρμακα, θα καταστρέψουμε τους μικρούς αγρότες, για τους οποίους ε, μίλησε η Λίδια, γιατί δεν έχουν ούτε τα χρήματα να, το, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, γιατί δεν είναι και βιώσιμος. Εμείς θα πρέπει να προστατεύουμε το έδαφος. Ε, θα πρέπει να προστατεύουμε τη βιοπικιλότητα στο έδαφος, γιατί τα χημικά και τα φυτοφάρματα καταστρέφουν και το χώμα, δεν καταστρέφουν μόνο τα ζυζάνια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα για αγροοικολογικές καλλιέργειες ε, και ε, ε, υπάρχει και επίσης πολύ μεγάλη γνώση αυτοχθόνων λαών και γεωργών με πατροπαράδοτες μεθόδους που ακολουθούνται εδώ και αιώνες. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Αν πάτε στην Αφρική, στην Υπεθρό, θα δείτε ότι ακριβώς αυτοί οι μικροί αγρότες παράγουν τρόφιμα. Τα 60% των τροφίμων παράγονται από αγρότες που έχουν λιγότερο από 2 εκτάρια. Αυτούς λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δική τους γνώση, τις δικές τους μεθόδους και να βρούμε και μεθόδους που να μπορούν ήδη να υπομισθούν οικονομικά. Ευχαριστώ. Η κυρία um, Ευχαριστώ. Χτες, Πρόεδρε, ήμουνα σε ένα γεύμα και συζητήσαμε εκεί ότι δεν κάνουμε αρκετά για την πείνα στον κόσμο και για τον υποσυτισμό θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχουν γίνει πάντω βήματα πρόοδου, μόνο που απομένουν πολλά ακόμα για να γίνουν. Πολύ ενδιαφέροντα τόσο όσα μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο που κράτησα είναι ότι θα πρέπει να ε, δούμε τι στοιχεία, τι ενδείξει υπάρχουν και από την άλλη μεριά είναι το πώ θα γίνουν περισσότερα. Θα πρέπει ε, ναι, να λάβουμε υπόψη το θέμα του ότι σύμβουλοι χρειάζονται περισσότερε αναπτυσσόμενε χώρε εκεί και σε επίπεδο ακόμα γεωργικής ε, εκμετάλλευσης ε, χρειάζονται συμβουλή και όχι στον ανεπτυγμένο κόσμο. Αυτό θα πρέπει να θεωρήσει μπούσουλα η ε, Κομισιόν. Αύξηση επίσης παραγωγής τροφίμων, αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, γιατί έχουμε από την παραγωγή του, των τροφίμων από τη μία μεριά βέβαια παραγωγή βλαπτικών αερίων, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή αυτών των τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλα τα τρόφιμα που απορρίπτουν, γίνονται σκουπίδια και δεν χρησιμοποιούμε και άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ήδη κάποια απτά αποτελέσματα και ότι οι πρωτοβουλίες μας θα μας δώσουν δυνατότητα να βελτιώσουμε την κατάσταση ούτως ώστε η πρόσβαση ε, στα είδη διατροφή να γίνει μια πραγματικότητα για τον κόσμο. Να δούμε τι θα γίνει και με τον υποσυντισμό. γιατί όσον αφορά τα παιδιά αυτό είναι κάτι που τα πλήσει και το πληρώνουν όλου στη ζωή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Χόισλεγκ. Ευχαριστώ. Πολλά είναι τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη συζήτηση αυτή και με εκπλήσει που υπάρχουν κάποιοι βουλευτέ ε, που, που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Εντάξει, τι να τους κάνουμε αυτούς. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη γεωργία σε συνεργασία με την αναπτυξιακή συνεργασία ακριβώς. Εμείς που ασχολούμαστε με τη γεωργία, αν δούμε τι κάνει η Ευρώπη στην αναπτυξιακή ε, συνεργασία και βοήθεια είναι και άλλα χημικά και άλλα λιπάσματα και άλλα φυτοφάρμακα και όχι προσαρμοσμένα συστήματα. Δεν μπορούμε τα δικά μας μοντέλα να τα αντιγράψουμε μόνο με γενετική τεχνολογία και χημεία θα λύσουμε το πρόβλημα και θα έχουμε και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία. Χρειαζόμαστε νέα μοντέλα προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα, την εκάστοτε. Μιλάμε για την παγκόσμια διατροφή και θέλουμε το δικό μας μοντέλο να το μεταφέρουμε εκεί. Το 70% ε, των σιτηρών μας ε, γίνονται ζωοτροφές και 15 εκατομμύρια δίνει ο Επίτροπος για τη Γεωργία ε, για να κάνει διαφήμιση για να τρώμε λέει περισσότερο κρέας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ε, μιλήσαμε για μια Γεωργία κλιματικός ευφυή για να το συζητήσουμε αυτό γιατί καμιά φορά έχουμε ε, ε την εντύπωση ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη γλυφοζάτη και άλλες τέτοιες χημικές ουσίες για να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Δηλαδή να σταματήσουμε και να οργώνουμε ακόμα γιατί θα τα κάνει όλα η χημεία και τα φυτοφάρμακα. Και δεν πειράζει για το έδαφος και για το χώμα. Γίνεται συζήτηση για τα τρόφιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο που ωρεοποιούμε την κατάσταση και αντί να καλλιεργούμε δημητριακά ή ε, καλλιέργειες ε, για τρόφιμα, παίρνουμε φωτοβολταϊκά για παράδειγμα. Και μετά εισάγουμε ε, και σόγια και ζαχαροκάλαμο, ζάχαρη δηλαδή, που δεν είναι καθόλου για τρόφιμα ή για το ζαχαροκάλαμο το χρησιμοποιούν ως καλλιέργεια για να παράγουν καύσιμα για τα αυτοκίνητα νέες τεχνολογίες χρειάζονται προσαρμοσμένες σε συνεργασία με ε, ντόπιου κάθε φορά. Δεν μπορούμε να γράψουμε το δικό μας μοντέλο και να το φυτέψουμε παντού. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ε, Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το ζήτημα αυτό. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε όταν κάποιος παράγει είναι να εξασφαλίσει ότι δεν πετάει, δεν το 30% της παραγωγής όταν λέμε να παράγουμε περισσότερα, ε, πρώτα καλύτερα να σταματήσουμε να σπαταλάμε. Είναι ένα μεγάλο μέρο του προβλήματο αυτό. Υπάρχει ένα άλλο μέρο του προβλήματο όμω που οι άνθρωποι έχουν τρόφιμα, αλλά αυτοί του ανθρώπου του πυροβολούν. Και τα όπλα αυτά παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να, να, να καλλιεργήσουν τη γη του γιατί του βομβαρδίζουν. Είναι και αυτό ένα μεγάλο μέρο του προβλήματο. Ένα άλλο μέρο του προβλήματο είναι ότι δεν κλείνουμε τον κύκλο δεν υπάρχει απορρόφηση των ε, απορριμμάτων. Δεν μειώνουμε τη χρήση λιπασμάτων. Και, έτσι ζημιώνουμε ακόμα περισσότερο περιβάλλον. Αυτό που χρειάζεται, αυτό που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, είναι το αριστερό και το δεξί χέρι να είμαστε βέβαιοι ότι είναι συνδεμένα με το ίδιο σώμα. Διότι αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ, λαμβάνει η χώρα και ταυτόχρονα στο παρασκήνιο Έχουμε τη ΣΕΤΑ, έχουμε το TTIP, έχουμε το Μερκοσούρ. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αλλά τι νόημα έχει να έχουμε πλοία τα οποία έχουν τα ίδια προϊόντα και το ένα μετα, το μεταφέρει από το α στο β, άλλο από το β στο α. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιοφυΐα για να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ακόμα και χώρες όπως η Ιρλανδία, που εκποφελούνται από αυτό, ας πούμε. Δεν είμαστε καν κυρίαρχοι σε ό,τι αφορά το τρόφιμά μας. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το ΣΕΤΑ, η TTIP, το Μερκοσούρ. Μα τι κάνουμε. Και τι τα συζητάμε αυτά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελαέ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά αυτό το θέμα είναι συναρπαστικό. Είπαν οι συνάδελφοι πάρα πολλά. Να μην ξεχνούμε επίση ότι η πείνα και ο υποσυτισμός δεν είναι φαινόμενο μόνο εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σοβούν και εδώ στην κοινή αγορά. Το είπε πριν από λίγο ο κύριος Φλάνεγκαν και το πρόβλημα τις ε, διασπάθηση των τροφίμων δεν είναι μόνο κάτι κακό για την παραγωγή, αλλά ε, γίνεται μόνο στην επίπεδο του παραγωγής, γίνεται και από τον κάθε καταναλωτή, από το ψυγείο του. Να, έτσι γίνεται από την ε, κοινωνία της κατανάλωσης. Αγοράζουμε πολύ περισσότερο από τις ανάγκες μας, οπότε στη συνέχεια πετάμε αυτά που περισσεύουν. Το ίδιο γίνεται και με τα τρόφιμα. Οπότε είχαμε και αυτή την, ε, τον εορτασμό στο Κοινοβούλιο για την οικονομία της αλληλεγγύης, την κυκλική και οικολογική και οπότε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντική πρόκληση, σημαντικό πρόβλημα να λύσουμε το πώς θα θρέψουμε αυτή την, ανθρωπότητα που να είναι πιο πολύ άρεθμη. Ευχαριστούμε κύριος Έκλε, πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Παγκόσμια Μέρα Διατροφής και η σημερινή συζήτηση είναι υπό την επικεφαλίδα «Αλλάζει το κλίμα, θα πρέπει να αλλάξει και η γεωργία και η διατροφή». Σωστό. Αλλά ε, δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρω, κάποιοι συνάδελφοι θα θυμώνται την πρώτη μου ομιλία εδώ στην Επιτροπή που είχα πει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι στη γεωργία Αλλιώς θα χάσουμε το κλίμα, θα πρέπει να μειωθούν οι μεγάλες ε, κτηνοτροφικές ε, μονάδες. Ε, με χλέβασαν, μου είπαν ότι είμαι βίγκαν είμαι και πραγματικά το συζητάμε αλλά όχι αρκετά. Και θέλω να πω ότι έχει δίκιο ο Χόισλινγκ. Είναι δυνατόν ένας Ευρωπαίος Επίτροπος όταν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και τάσεις στην κοινωνία να πετάει 15 ε, εκατομμύρια ευρώ για μια διαφήμιση για να αυξηθεί η κατανάλωση κρέατος και μάλιστα βοήου κρέατος. Μεθάνιο, σε τεράστιες ποσότητες βάζουν τα βοηδή. Κάθε μέρα να μετρήσουμε τι φεύγει στην ατμόσφαιρα. Και τι λένε τα προγνωστικά, 320 εκατομμύρια τόνους κρέας παράγουμε και το 2050 πάνω από 600 εκατομμύρια τόνους είναι οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις. Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Και πάνω από τη μισή καλλιέργεια των σιτηρών στον κόσμο είναι για ε, ζωοτροφές και πάνω από 90% της όγιας είναι για ζωοτροφές και θέλουμε να κάνουμε και εκστρατεία για να τρώει ο κόσμος βόλιο κρέας. Αυτά τα πράγματα είναι φρικιαστικά και δεν μπορώ παρά να σας κάνω την εξής μια στιγμή κύριε Λαβία, μια συμβουλή. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό για να ε, μιλήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάψουμε τον κύριο Χόγκαν και να τον αλλάξουμε με ένα πιο φιλόδοξο επίτροπο για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να μην πεινάει και τη γεωργία παγκοσμίω. Ευχαριστώ κυρία Τόρης Μαρτίνες. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που επιτέλους αποφασίσαμε σε επίπεδο του Κοινοβουλίου να μιλήσουμε για τις απαραίτητες αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα γεωργίας και σύντησης. Δεν έγινε αναφορά πουθενά σε αυτό στη συμφωνία του των Παρισίων. Ελπίζω λοιπόν αυτή η συζήτηση ε, να αποτυπωθεί κάπως στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Μαρακές και εκεί η Ευρώπη να προσεγγίσει αυτή την αναγκαιότητα να προωθηθεί η οικολογική γεωργία και ε, τα μικρά κυκλώματα παραγωγής. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να φάει βιώσιμα, ισότιμα και θα μειώσουμε και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει ένα μικρό μέρος της δημόσιας ενίσχυσης στον τομέα της έρευνας να του αφιερώσουμε εκεί και να μην τα αφιερώνουμε ε, στα μεταλλαγμένα. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, το λέει και η ΦΑΟ, το λέει και η Παγκόσμια Τράπεζα ακόμα. Αυτό όμω πρέπει να είναι σαφέ είναι ότι δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε αλλαγή στη γεωργία και στη διατροφή, να μιλάμε για ε, κυριαρχία στη διατροφή, ενώ από την πίσω πόρτα προσπαθούμε να φτάσουμε σε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών όπω το ΣΕΤΑ και το TTIP που πάνε προ την αντίθετη κατεύθυνση. Θα πρέπει να φανούμε εδώ ειλικρινεί. Όχι μόνο λόγια αυτοί που μας έβαλαν σε αυτό το, το νίκο πρέπει να τους τιμήσουμε, να τιμήσουμε την ψήφο τους. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε τις, τα σχόλια των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια σύντομη, σύντομη αντίδραση παρακαλώ από πλευράς ΦΑΟ. Thank you very much to the three chairs and the members again for for this opportunity. Σας ευχαριστούμε την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ τους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους που έδειξαν το ότι πρέπει να έχουμε την ευκαιρία για να διορθώσουμε τα πράγματα αλλά είναι και άλλα σημαντικά που ελέγχθησαν ότι δηλαδή έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και ότι επομένως θα πρέπει αυτό να μας ενθαρρύνει να κάνουμε την διαφορά, να συνεργαστούμε. Παγκόσμιο να υποστηρίξουμε τις χώρες και να δράσουμε επί τόπο. Οπότε βεβαίω και θα λάβω υπόψη όλα όσα σήμερα άκουσα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα. Θα πρέπει επίσης να βοηθούμε τις χώρες για να υλοποιήσουν τις ε, στρατηγίες που έχουν χαράξει και τις άλλες δράσεις. Φάνηκε από τα όσα ακούσαμε σήμερα ότι είναι πολύ σημαντικό να ενεργούμε με τα λόγου γνώσεως και να δούμε και να καταλάβουμε η κάθε προσέγγιση τι υπέρ και τι κατά έχει, τι είναι το πιο δόκιμο στο κάθε ε, πλαίσιο μέσα στο οποίο βρούμε στις συνθήκες που ζούμε. Θα συνεργαστούμε με την ΤΕΦΚΟ και στο μέλλον για να εξευρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ο πρώτος ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτό το, το κομμάτι της συνεδρίασης και θα λάβει την ε, σκητάλη ο κύριος Σικέρσκι. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε από κοινού με τον ΦΑΟ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εμείς, τα μέλη των τριών κοινοβουλευτικών ε, επιτροπών, περιβάλλοντος, ανάπτυξης και γεωργίας. Να δούμε πώς θα υπάρχει επισυντισμός για όλο τον κόσμο. Και αυτά έχουν άμεση σχέση βέβαια με την ε, Διεθνή Μέρα Επισυντισμού. Πρόκειται για προβληματική που κρατάει πολύ καιρό. Όπως είπατε, έχουμε 800 εκατομμύρια που έχουν πρόβλημα υποσυντισμού και πείνας. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα πιο συγκεκριμένα. Το τι πάει να πει φαγητό μπορεί να σας το εξηγήσει πολύ καλά κάποιος ο οποίος πεινάει. Αυτά άλλωστε τα έζησε ο κόσμος και στον πόλεμο και με τα πολεμικά. Αλλά και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια στην Ευρώπη που απειλούνται από το έλλειμμα που υπάρχει για στον επισητισμό στην κατά τα άλλα πλούσια Ευρώπη. Μιλούμε για 80 εκατομμύρια στην Ευρώπη που έχουν πληγεί από αυτό το πρόβλημα στον επισητισμό, στην ανεπάρκεια. Οπότε η κοινή γεωργική πολιτική ήταν γι' αυτό το λόγο η πρώτη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που χαράχθηκε. Εξελίχθηκε. Μετά συνδέθηκε περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον. Αλλά νομίζω ότι η γεωργία μας δεν πρέπει να είναι πιο φιλική προς τη φύση και το περιβάλλον. Βέβαια σήμερα δεν συζητούμε, τούτο συζητούμε το τι γίνεται με την αλλαγή του κλίματο. Πολύ σημαντικό και αυτό σε σχέση με τη γεωργία. Τη γεωργία δημιουργεί βλαπτικέ εκπομπέ, όμω και απορροφά ε, εκπομπέ. Απορροφά διοξίδιο του άνθρακο. Έχουμε την φωτοσύνθεση. Και άρα η γεωργία είναι πηγή καλών για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Στην τελευταία μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε αυτό το greening, το πρασίνισμα της πολιτικής να γίνει πιο φιλική για το περιβάλλον και για τη φύση. Και η οργία και τα δάση ε, όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος βοηθούν πάρα πολύ, περιορίζουν τις βλαβικές συνέπειες. Γι' αυτό μιλήσαμε για την διακράτηση, κατακράτηση του διοξιδίου και επίσης είναι και πολύ σημαντικό, σημαντική κλάδη ε, για τη διαχείριση του, του νερού, των υδάτινων πόρων. Και η πέθρος βέβαια είναι πολύ σημαντική γιατί από εκεί ξεκινά η υπόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε ότι θέλουμε να αναπτυχθούν οι μεταφορές, είπαμε ότι θέλουμε τα είδη διατροφής, να προέρχονται εκατομμύρια εξεργασίας από τα γεωργικά προϊόντα και ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την παγκόσμια αγορά. Αλλά έχουμε και εξωγενείς παράγοντες, εξωγενείς μεταβλητές. Έχουμε τις διεθνείς συμφωνίες. Πρόεδρε, δεν θα με άλλο. Μην ξεχνούμε ότι εξωτερικό εμπόριο δεν σημαίνει μόνο ε, ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων. Δεν πρόκειται μόνο για πόλεις, είναι ανταλλαγή κυρίως. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε εις βάθος, να τα μελετήσουμε καλύτερα. Θέλουμε να έχουμε πλέον εκτήματα, αλλά αυτό να στηρίζεται σε συνεργασία, σε εταιρική σχέση και να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι σε όλη την διαδρομή. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την ιδιωτική πολιτική και την ε, παραγωγή ειδών διατροφή. Νομίζω ότι στο μέλλον θα είναι τα πράγματα πιο καλά για το περιβάλλον, θα είναι πιο φιλική η παραγωγή στο περιβάλλον. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε σήμερα, του στόχους, τι προκλήσεις, ε, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί ήδη έχουμε καταφέρει αρκετά. Έχουμε κάνει πολλά που να μα κάνουν ε, υπερήφανου. Μην ξεχνούμε όσο έχουμε πετύχει. Έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή γεωργική πολιτική. Είναι ε, ό,τι καλύτερο έχει κάνει. Πρέπει να συνεχίσει να έχει προτεραιότητα βέβαια η γεωργική πολιτική στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σικέρσκη, λέει ο πρόεδρο. Όλου σα ευχαριστώ για αυτήν την ε, κοινή συνεδρίαση των ε, τριών ε, επιτροπών συνάντηση με τον ΦΑΟ εδώ. Θα κάνουμε μια διακοπή στην συνεδρίαση, ώστε να μπορεί να αποχωρήσει όποιο θέλει. Και σε δύο λεπτά συνεχίζουμε. Θα έρθει ο επίτροπο κ. Ναι. Μπούλτ ή η Επιτροπή κ. Μπούλτ για την υπόλοιπη συνάντηση.